η συζήτηση σχετικά με τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης τώρα είναι ήδη διαθέσιμα εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια στα πρακτικά αυτά συνεπώς θεωρούνται δεκτά η μερίσια διάταξη τώρα μας οδηγεί σε ερωτήσεις την παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζετε τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τη συγκεκριμένη μορφή συζήτησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα